Καλησπέρα, συνάδελφοι. Συνεχίζουμε. Τη συνεδρία στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι ερωτήσεις προς το Συμβούλιο. Καλωσορίζω εδώ τον Υπουργό εκ μέρους της Βελγικής Προεδρίας. Η πρώτη ερώτηση είναι η ερώτηση της κυρίας ε, Βίνκερ Φλούτσε σχετικά με άτομα με αναπηρία και τη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Κύριε Υπουργέ, όταν είσαστε έτοιμος, παρακαλώ να απαντήσετε. Madame Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβούλιο δίνει μεγάλη σημασία